Λοιπόν, να αρχίσει λοιπόν, ξανά η συνεδρία. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά γιατί να αρχίσουμε συνεδρίαση χωρίς να είναι παρόντα τα μέλη μας. Περνούμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η εβδομάδα κινητικότητας και η σχετική μήνυα ακρόαση. Όπως γνωρίζετε ε, η συνεδρίαση είναι μεσούς της ε, εβδομάδας αυτής και είναι και δεκαετία από την αρχή της πρωτοβουλίας και είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα αηφόρου κινητικότητας της πόλης ε, πέρα από σύνορα. Τέσσερις ομιλητές έχουμε μαζί με την Ισαμπέλ Τυρό που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Αντρέη Κολόμπο που είναι σύμβουλος κινητικότητας και ε, μεταφορών της, ε, του Δήμου της Μπολόνια, τον κύριο Πίτερ Βαντσέβαντ που είναι επικεφαλής ε, της αντίστοιχης υπηρεσίας της πόλης της Γάνδη και τον αντιδήμαρχο του Δήμου του Βίλνιους από τη Λιθουανία. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Τζιρό, αφού καλωσορίσω τους προσκεκλημένους, να πει δύο λόγια για δέκα λεπτά και μετά δέκα λεπτά κάθε ε, εμπειρογνώμων και μετά ερωτήσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε όλοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις πόλεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και ήρθαν στην Επιτροπή Μεταφορών για να μας δείξουν ε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα. Και τις EuroCities θέλω να ευχαριστήσω για τις προτάσεις τους αυτές. Ε, βεβαίως είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό, να δούμε τι πρόοδοι έχουν επιτευχθεί σε κάποιες πόλεις. Τρεις σήμερα θα συναντήσουμε και είναι πολύ πιο ενδιαφέρον που εκτός από αυτές τις πρωτοπόρες όπως θέλουν να είναι πόλεις και θα δούμε με ποιο τρόπο το έκαναν, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές πόλεις που είναι σε κάποιο τέλμα, δεν μπορούν να βγουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν τα βγάζουν πέρα, δεν βρίσκουν τον τρόπο, τους μοχλούς, τους μηχανισμούς για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Για διάφορους λόγους, αδράνεια, υποδομές, το παρελθόν, η δομή της πόλης, το γεγονός ότι είναι κεντρική, περιφερειακή, ότι έχει ε, καθημερινή κίνηση ή όχι. Κάθε πόλη έχει την ιστορία της. Αλλά πολλές ε, πόλεις έχουν πρόβλημα να ε, φύγουν προς τα μπρος. Πριν από κάποιες δεκαετίες κυριαρχούσε το αυτοκίνητο. Σήμερα έχουμε κάποιες προτάσεις και θα τις ακούσουμε για να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για να έχουν πιο αηφόρο, πιο ήπια και εναλλακτική κινητικότητα. Είμαι βέβαιη ότι θα απαντήσουν στο ερώτημα οι εμπειρογνώμονες τι μπορεί να κάνει επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να βοηθήσει ε, όταν βέβαια είμαστε στα χωράφια της επικουρικότητας. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις, τι μοχλούς πίεσης έχουμε και δράσεις και οι κύριοι εκπρόσωποι των πόλεων αυτών, ποια είναι η άποψή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθέτησε μετά από πολλά χρόνια για τα δικαιώματα των επιβατών που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα μπορούσε ε, να νομοθετήσει και για τους χρήστες των ε, αστικών συγκοινωνιών ε, σε πόλεις που κυριαρχεί ακόμα το αυτοκίνητο για να έχουμε καλύτερη και πιο άνετη ζωή όχι μόνο για τους πολίτες της πόλης μας αλλά να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη οικονομική ελκυστικότητα για τις πόλεις που θα έχουν απελευθερωθεί από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και όπου θα έχει μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας. Αυτό έγινε με το σύμφωνο των δημάρχων. Ξέρετε ότι στα πλαίσια των προγραμμάτων για την ενέργεια ήταν αυτό το σχέδιο, το σύμφωνο των δημάρχων. Ε, θα μπορούσε να γίνει και μια συνέλευση αντίστοιχη των δημάρχων για να ε, δώσουν προτάσεις ε, στους δημάρχους και σερετούς των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλων για να μπορέσουν να κινηθούν προς τις αστικές συγκοινωνίες και την κινητικότητα καλύτερα που να είναι πιο αποτελεσματική, πιο αποδεκτή και να είναι και οι πόλεις πιο ελκυστικές. Αυτά ως ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα τονίσετε τα θέματα, τα βήματα που κάνετε εσείς και τι περιμένετε από μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Ο πρώτος ομιλητή, ο κ. Κάρλο Καρλίνη, και ζητώ συγγνώμη που είπα λάθο το όνομά σα, Είχα το είχα λάθος γραμμένο. Είναι από την πόλη της Μπολόνιας. Θα ξεκινήσει την παρουσίασή του πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ο μιλητής, και την Αντιπρόεδρο. Ανήκω στο Δήμο της ε, Μπολόνιας, ασχολούμαι με την κινητικότητα. Ε, είμαι δημοτικό Σύμβουλος και ασχολούμαι και με δράσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα και σχετίζονται και με τον προϋπολογισμό. Στη σημερινή παρουσία θα προσπαθήσω σε λίγα λεπτά να σας πω ποιες είναι οι στρατηγικές που προωθούμε και προωθήσαμε τα τελευταία χρόνια υπέρ της ε, βιώσιμης κινητικότητας. Θα εστιαστώ κυρίως στο τι καταφέραμε και κυρίως χάρη στην ε, συμμετοχή και συνεργασία της Ευρώπης. Καταρχάς, ε, δύο λόγια την Πολόνια. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ιταλίας, είναι μεσαία πόλη, περίπου 400.000 κατοίκους έχει, αλλά όμως είναι σημαντικός κόμβος ανταλλαγής ε, και συμμετέχει σε όλες τις εθνικές ροές. Από εκεί περνάνε, από την Πολόνια, οι μεγάλες, ε, οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι και οι μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές της Ιταλίας. Επίσης, επίσης ως πόλη παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις ροές και στις ανταλλαγές ε, των μεσογειακών πόλεων πάρα, πάρα πολλές κινήσεις, ροές ε, ε, παρατηρούνται. Έχουμε περίπου 2 ε, εκατομμύρια άτομα που μετακινούνται. Περίπου το 50% μπαίνει προς την πόλη και το υπόλοιπο είτε μετακινείται, εκτός πόλης δηλαδή, είτε περνάει από την Μπολόνια και να πάει κάπου αλλού προς, τα, προς άλλη κατεύθυνση. Αυτά τα δεδομένα, η θέση μας, το γεγονός ότι είμαστε μια μητροπολιτική πόλη για την Ιταλία, μας φέρνει σε επαφή και με άλλες Ιταλικές πόλεις και ευρωπαϊκές πόλεις σε ό,τι αφορά την τις μεταφορές, έχουμε προβλήματα βεβαίως κυκλοφοριακής συμφόρησης και βεβαίως είχαμε προβλήματα ρήμα, ε, ρήπανσης. Ξέρετε βεβαίως ότι ο βοράς της Ιταλίας, ε, η κοιλάδα του Πάδου, ε, γνώρισε πολλά προβλήματα με, λεπτές, ε, με λεπτά εωρήματα σκόνης. Ε, είχαμε προβλήματα ρήπανσης δηλαδή. Ε, στο παρελθόν, λοιπόν, απτύξαμε μια στρατηγική για να περιορίσουμε αυτούς τους ρήπους, ε, αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις ε, και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε δράσεις υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας. Ε, γκρίναμε, λοιπόν, ένα σχέδιο το 2007 για τη διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας ε, που υιοθετήθηκε και χάρη στην στενή συνεργασία με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, συμμετείχαμε στο EuroCities βεβαίως και συμμετείχαμε και στο, στην ανάπτυξη του προγράμματος Μιμόσας, στα πλαίσια του προγράμματος Τσιβιτάς Μιμόζα. Ε, Εδώ και 12 χρόνια συμμετέχουμε και στην Ευρωπαϊκή Βδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας. Και μάλιστα αυτές τις μέρες είναι εξελίξη. Τώρα, το πρόγραμμα Μιμόζα. Βλέπετε ποιοι είναι οι εταίροι μας. Ε, η Μπολόνια είναι ο συντονιστή του προγράμματο αυτού και συμμετέχει και η Ουτρέχτη, το Γκτάνσκ, το Τάλιν και το Φουντσάλ. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για 70 μέτρα. Από αυτά 18 αφορούν την κοινότητα της Μπολόνιας, δήμο καλύτερα στα ελληνικά της Μπολόνιας. Είχαμε διάφορους ε, τοπικούς ε, φορείς και εταίρους ε, από την περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια και υπάρχει και ο φορέας που διαχειρίζεται στην Ιταλία τις αστικές συγκοινωνίες, τις δημόσιες συγκοινωνίες. Η δράση μέσω του Μιμόζα μας έδωσε διάφορα ωφέλη. Το πρώτο είναι ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρήματα. Είχαμε στη διάθεσή μας χρήματα δηλαδή. Θα σας εξηγήσω αργότερα πώς χρησιμοποίησαμε αυτά τα λεφτά που μας δόθηκαν χάρη σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότηση στο Μιμόζα. Ε, ήταν επίσης σημαντικό το ότι συμμετείχαμε σε αυτό το πρόγραμμα για να προωθήσουμε μέτρα ε, συμμετοχής των πολιτών και να δημιουργήσουμε κάποια εργαλεία για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων και να ανταλλάξουμε και απόψεις, ούτω ώστε να εισαγάγουμε και να εξάγουμε ε, τις θετικέ εμπειρίε μας στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για την βιώσιμη κινητικότητα. Πολύ σύντομα τώρα θα σας δείξω κάποια από τα μέτρα τα οποία προωθήσαμε και χάρη στην σημαντική συνεισφορά του προγράμματος Τσιβιτάς Μιμόζα. Ε, βελτιώσαμε καταρχάς και τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα οχήματα δηλαδή, αλλά και τα ιδιωτικά. Ε, είχαμε καινοτόμα μέσα με τους σούπερ πυκνοτές που βελτιώσαμε τρομερά ε, την εξοικονόμηση ενέργειας, μειώσαμε τους ρήπους, ε, προωθήσαμε ε, επίσης ιδιωτικές ροές, δηλαδή ιδιωτικέ, ε, ιδιωτικά οχήματα. Ε, δώσαμε κίνητρα για να απτυχθούν Ε, γιοταχή, τα οποία όμως χρησιμοποιούν ε, συστήματα λιγότερο ρηπογόνα. Σήμερα στην Πολώνια, ας πούμε, ε, πάνω από 16% ε, τροφοδοτείται με υγραέριο και με άλλα μέσα. Επίσης, δημιουργήσαμε αυτό το car sharing, επιμερισμένα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα που τα χρησιμοποιούν πολύ και έχουμε και συστήματα ελέγχου της στάθμευσης. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν μερικές φορές χώρες στάθμευσης και χρησιμοποιούνται λάθος. Ε, δεν προ... Συχνά δεν τα χρησιμοποιούν αυτοί που θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούν. Εμεί τι κάνουμε λοιπόν, έχουμε διάφορου τρόπου για να κλείνουμε αυτού του χώρου στάθμευση, διάφορα εμπόδια α πούμε, ούτω ώστε να χρησιμοποιούνται ε, από αυτά αυτού που συμμετέχουν στο car sharing. Μια άλλη δραστηριότητα είναι ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ε, χώρων στάθμευσης. Μπορεί κανείς να παρκάρει δωρεάν, εφόσον έχει το εισιτήριό του ε, για το λεωφορείο ή για οποιαδήποτε δημόσιο μέσο μεταφοράς. Χάρη στο Μιμόζα ε, βελτιώσαμε δύο από αυτούς τους χώρους στάθμευσης που είχαμε, δύο από αυτά πάρκινγκ. Επίσης άλλες ουσιαστικές δραστηριότητες είναι οι δράσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ε, το θέμα των τροχαίων και των θανατηφόρων τροχαίων ε, για την Ιταλία είναι πραγματικά μάστιγα. Είναι πολύ σημαντικ... Ήταν πολύ σημαντικό ο αριθμό και είναι σημαντικό ο αριθμό. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε μια σειρά δράσεων. Φερρυπίν, α πούμε, βελτιώσαμε την ασφάλεια κάποιων σταυροδρομιών. Και επίση ε, βάλαμε σε διάφορε σημεία τη πόλη σε όρια ταχύτητα 30 χιλιόμετρα, ούτω ώστε να περιορίσουμε την χρήση των γεωταχή των κλασικών γεωταχή. Επίσης, θεωρούμε για το θέμα της ασφάλειας ε, πολύ σημαντικό την συμμετοχή των πολιτών και των παιδιών. Προηγουμένω μιλούσα για τους, μιλούσατε μάλλον για τα, τους αδύναμους χρήστες. Σίγουρα τα παιδάκια είναι από τους πιο αδύναμους χρήστες. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε δράσεις για την ασφάλεια των παιδιών και των, και γονιών τους όμως. Χθε, ας πούμε, στην Πολόνια ξεκίνησε η σχολική χρονιά και έχουμε 7 συστήματα, θα έλεγα, πεζολεοφορίων. Δηλαδή, ε, κάποιο βοηθάει τα παιδιά, τα, τα, τα, τα περπατάει ουσιαστικά ως το σχολείο χωρίς να χρησιμοποιείται κανένα μέσο μεταφοράς. Επίσης, έχουμε έξυπνα συστήματα υπέρ της κινητικότητα. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ και χρηματοδοτούνται μέσω του Μιμόζα. Ένα σύστημα, παραδείγματο χάρη, για τον ε, έλεγχο της, ε, του διπλοπαρκαρίσματος μέσω ενός ανοιχνευτή του Σκάουτ. Επίσης έχουμε το STARS, ελέγχουμε τα φανάρια δηλαδή και κάτω-κάτω βλέπετε ε, στα Σταυροδόνια εκεί που βάλαμε αυτό, τα, αυτά τα συστήματα έχουμε μειώσει κατά το 50% τα ατυχήματα. Χάρη σε αυτές τις καινοτομίες το 2010 αναγνωρίστηκε ότι η Μπολόνια είναι έκανε πολλές προσπάθειες και της δόθηκε βραβείο στην τελετή του προγράμματος ΣΥΒΙΤΑΣ. Επίσης, για την τεχνολογία που έχουμε, ε, δημιουργήσαμε ζώνες, μεγάλες, ευρείες ζώνες ε, πεζόδρομων, γύρω από το Πανεπιστήμιο Φαραδί. Εκεί περιορίσαμε την χρήση των γεωταχή και των ε, τετράτροχων και των δίτροχων, δηλαδή και των μοτοσυκλετών. Ε, μειώθηκε κατά 70%. Και ουσιαστικά ξαναδώσαμε δηλαδή την περιοχή αυτή, την ξαναχαρίσαμε ε, στους πιο αδύναμους χρήστες ε, και στους πεζούς. Να κάποιες φωτογραφίες εδώ που βλέπετε, που βλέπετε πώς είναι η σημερινή κατάσταση με αυτές τις πρωτοβουλίες, με πρωτοβουλίες που οργανώνονται χάρη σε αυτόν τον χώρο που ξαναανακτήσαμε από τα αυτοκίνητα. άλλη δράση στα πλαίσια του Μιμόζα. Από το 2002 συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, ε, προωθούμε πάρα πολλές δράσεις και αυτές τις μέρες μάλιστα προωθούμε διάφορες. Σημαντικό είναι να εμπλακούν και οι πολίτες εδώ. Εδώ τονίζω την δραστηριότητα προωθήσαμε πέρυσι το 2011, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο ε, το οποίο είχε αρχίσει να δουλεύει τον, λίγους μήνες πριν, αποφάσισε τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας να τις κάνει πεζόδρομους. Ε, και το Σαββατοκύριακο δεν κυκλοφορεί κανένα όχημα εκεί πέρα. Μόνο ε, ποδηλάτες και πεζοί. 60.000 άτομα πήγαν στο κέντρο, λοιπόν, της, πήγαν στο κέντρο της Μπολόνια, στο ιστορικό κέντρο, όπου ήταν ε, πεζοδρομημένοι και το Φεβρουάριο που μας πέρασε αναγνωριστήκαμε ως η καλύτερη πόλη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δομάδας για την Κινητικότητα που οργανώθηκε το 2011. Στο μεταξύ κάναμε και άλλους πειραματισμούς. Από το Μάιο του 2012 αυτό το μέτρο το προωθούμε ε, τακτικά κάθε Σαββατοκύριακο δηλαδή, το κέντρο, το ιστορικό κέντρο της Μπολόνιας ε, κλείνει εντελώ τα οχήματα και γίνεται, ε, το δίνουμε ας πούμε στους πεζούς και στους ε, ποδηλάτες. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά για να αναπτύξουμε περαιτέρω τις αστικές συγκοινωνίες, θα πρέπει να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την οδική ασφάλεια. Η βοήθεια και η συνεργασία των εταίρων, παλιών και καινούριων, Ευρωπαίων, ε, είναι πολύ σημαντική. Ε, ετοιμάζουμε ένα σχέδιο που λέγεται το νέο κέντρο. Στις 13 ε, Οκτωβρίου θα γίνει μια μεγάλη εθνική πρωτοβουλία που σκοπό έχει να προωθήσει και να απλώσει τους πεζόδρομους. Και παρότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μας είναι δεινή, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε ψηλά στην ημερησία διάταξη το θέμα αυτό της βιώσιμης κινητικότητας, ούτως ώστε να προωθήσουμε και την κινητικότητα και την χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς. Είναι σημαντικό αυτό για να βελτιωθεί και η ζωή στις πόλεις μας και η ζωή των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Very Ευχαριστώ κύριε Καλίνη. Από το Δήμο της Γάνδης τώρα, επικεφαλής ε, της αντίστοιχης εταιρείας στη Γάνδη, ο κύριος Βανσενεβάντ. Ελπίζω να μην κατακρεώρησα το όνομά σας. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, as my colleague... Καλησπέρα. Όπως και ο συνάδελφός μου από την Πολώνια θα σας μιλήσω για τις εμπειρίες μας στο πλαίσιο του προγράμματος Civitas και συγκεκριμένα του ε, προγράμματος ΕΛΑΝ. Είναι το πρόγραμμα στο οποίο ε, εμείς συμμετείχαμε, το αντίστοιχο με τη Μιμόζα. Η Γάνδη ήταν μία από τις γετικές πόλεις στις οποίες ε, συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΛΑΝ, ε, μαζί με τη Λιουμπλιάνα και το Ζάγκραπ και υπάρχουν και άλλες δύο πόλεις που συμμετέχουν στο πλαίσιο μαθητείας, το Πόρτο της Πορτογαλίας και το Μπρνό στην Τσεχία. Το πρόγραμμα διήρκησε τέσσερα χρόνια από το Σεπτέμβριο του 2008 και θα λήξει τον Οκτώβριο του 2012 η εταίροι στην Γάνδη, ε, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΑΝ, ήταν 7. Πρώτα απ' όλα φυσικά ε, ο ίδιος ο, ίδιος ο Δήμος της Γάνδης, η εταιρεία Ντελίνια, που είναι οι αστικές συγκοινωνίες, τα λεωφορεία, η φλαμανδική εταιρεία ε, οδικών μεταφορών, η Maxmobile, η Student and Mobilitate, η, οποία παρέχει υπηρεσίες για τους ποδηλάτες, η Κάμπιο και τέλος το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ΕΛΑΝ στην Γάνδη ανήλθε στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ και η επιχορήγηση ήταν 4,4 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός ε, επιμερίστηκε ως εξής, το 56% ήταν για την υλοποίηση του προγράμματος, κυρίως προσωπικό, καθώς επίσης και τις επενδύσεις. Ε, σε μεγάλο βαθμό επενδύσαμε στην έρευνα και την αξιολόγηση, το 19%. Η επικοινωνία, η εκπαίδευση και τα σεμινάρια ε, κάλυψαν το 19%. Είχαμε λοιπόν 24 μέτρα σε 8 κατηγορίες που καλύπτουν σαν για παράδειγμα την διαχείριση των αστικών ε, συγκοινωνιών ή και τους ιδιαίτερα ευάλωτους. Εστιάσαμε στην υλοποίηση των διαφόρων ιδεών. Δεν ήταν ο στόχος μας να δημιουργήσουμε υποδομές, αλλά στην ε, πραγματικότητα καταφέραμε να υλοποιήσουμε ιδέες που, καινοτόμες που ήδη υπήρχαν και ποτέ δεν μπορούσαμε να τις ε, κάνουμε πραγματικότητα. Χάρη στο πρόγραμμα Civitas καταφέραμε να τις υλοποιήσουμε και να εισάγουμε αυτά τα μέτρα στην πόλη. Στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου δεν μπορώ να καλύψω όλα τα μέτρα που υλοποιήσαμε, γι' αυτό θα αναφερθώ μόνο ορισμένα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τι αστικέ συγκοινωνίε, τι δημόσιε αστικέ συγκοινωνίε, η Delaney είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τι συγκοινωνίε στη Γάνδη και στο πλαίσιο του προγράμματος Σύβητας δημιούργησαν ένα σύστημα με το οποίο ε, μετρήσανε με πολύ μεγάλη ακρίβεια την ενέργεια που καταναλώνει ένα τραμ και ανακάλυψαν ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν το 20% αυτής της ενέργειας με μικρές ε, αλλαγές, αλλάζοντας μικρές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο ανοίγαν, άνοιγαν οι πόρτες. Ε, χανόταν πολύ μεγάλη ενέργεια θερμική όταν άνοιγαν οι πόρτες. Και ο τρόπος με τον οποίο εξοικονομήσαν ενέργεια είναι ότι σταματάει ο εξαιρισμός την ώρα που ανοίγει η πόρτα και με αυτές τις μικρές αλλαγές ε, μειώνεται κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας που έχει φυσικά και ως αποτέλεσμα μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό σε οικονομικούς όρους μεταφράζεται σε 200.000 ε, ευρώ το χρόνο για την Γάνδη. Επίσης, ε, στις επόμενες διαδικασίες λήψης προσφορών, στους επόμενους διαγωνισμούς συμπεριέλαβαν αυτές τις ιδέες. Ένα άλλο μέτρο απευθύνθηκε στους εφήβους, οι οποίοι όπως γνωρίζετε δεν είναι και πιο φρόνιμοι επιβάτες. Είχαμε δημιουργήσει ένα, μια ειδική εκστρατεία μέσω την, ε, προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ε, νέους για τις κινδύνους. Ε, είχαμε προσωμείωση για παράδειγμα ατυχημάτων σε περίπτωση που πιάσει φωτιά ένα λεωφορείο ή για να καταλάβουν πόσο Δύσκολο είναι κάποιο να ε, σβήσει ένα γκράφιτι που κάποιο μπορεί να έχει κάνει πάνω σε ένα λεωφορείο. Αποτέλεσμα, τέτοια περιστατικά μειώθηκαν κατά 53% στην πόλη μας. Οι ίδιες ιδέες και πάλι ε, δόθηκαν ε, και υλοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακαίνησης των σταθμών του τρένου, των σιδηροδρομικών σταθμών. Χάρη στο πρόγραμμα Civitas μπορέσαμε να εμπλέξουμε τους πολίτες με καινοτόμους τρόπους. Δώσαμε τη δυνατότητα στους πολίτες να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, μέσω του Civitas μπορέσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι συνήθω καταφέρνουμε. Τώρα στο θέμα της ε, διαχείριση της ε, κινητικότητας, είχαμε προγράμματα σε, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ξέρετε οι ε, έφηβοι είναι δύσκολο να πιστούν σε ζητήματα αηφόρου κινητικότητας, αλλά καταφέραμε μέσω διαγωνισμών να τους δώσουμε την δυνατότητα οι ίδιοι να προτείνουν ιδέες και καταφέραμε μέσω των προγραμμάτων να δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο μια ε, ε, πολύ ωραία, πολύ ωραία μικρή ταινία για τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επιβατών. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργήσαμε χώρους στάθμευσης ε, για τα ποδήλατα, είναι αρκετά τα ποδήλατα στη Γάνδη, Και ε, επίσης χρειάζεται και ένας τρόπος για να μπορεί κανείς να παρκάρει ε, καλά το ποδήλατό του όταν ε, το χρησιμοποιήσει στις καθημερινές του μετακινήσεις. Δημιουργήσαμε λοιπόν χώρου στάθμισης σαν αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Αυτό μας έδωσε εμπειρία την οποία τώρα ε, αξιοποιούμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και νέους χώρους στάθμευσης σε 20 ακόμα σημεία στην ε, πόλη και υπάρχει και μια μεγάλη λίστα αναμονής θέλουν ε, σε πολλά άλλα σημεία να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι στάθμευσης. Και πάλι δεν θα είχαμε μπορέσει να υλοποιήσουμε αυτό το έργο χωρί την βοήθεια του ΣΥΒΙΤΑΣ Επίση, καταφέραμε να διαδώσουμε, να συλλέξουμε και να διαδώσουμε τι πληροφορίε σε σχέση με τα ποδήλατα δημιουργήσαμε μια ειδική ιστοσελίδα και ε, μια ε, λειτουργικότητα αυτή τη ιστοσελίδα είναι ότι μπορεί κανείς να σχεδιάσει τη διαδρομή του. Ε, πολύ συχνά όσοι παίρνουν το ποδήλατό τους δεν γνωρίζουν τους ποδηλατόδρομους και έτσι μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορεί κανείς να ε, σχεδιάσει τη διαδρομή του και να αποφύγει τις συμφορήσεις, ή να αποφύγει τις γραμμές του τραμ ή να αποφύγει τους πολυσύχνες τους δρόμους. Κατά μέσο όρο 2.000 ε, διαδρομές το μήνα σχεδιάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδα. Επίσης το πρόγραμμα car sharing της ε, κοινή χρήση αυτοκινήτων έχει επεκταθεί μέσω του προγράμματος Σίβητας. Ε, εισαγάγαμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Επίσης απευθυνθήκαμε σε νέες ε, ομάδες προτείνοντάς τους να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για παράδειγμα σε εταιρείε, και πώς μπορούν αυτοί να, να το συνδυάσουν με το, σε υπηρεσίες της Κάμπιο. Έτσι καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη και ως αποτέλεσμα του προγράμματος car sharing ε, το, το πρόγραμμα μάλλον ε, η χρήση των αυτοκινήτων αυτών αυξήθηκε κατά 23%. Συμπερασματικά, μέσω του προγράμματος Civitas μπορέσαμε να μάθουμε νέα πράγματα. Είχαμε, ε, δημιουργήσαμε νέες διαδικασίες και νέα μεθοδολογία αξιολόγησης. Πάντα είχαμε δείκτες, αλλά τώρα χάρη στο πρόγραμμα του Civitas καταφέραμε να δημιουργήσουμε νέους τρόπους μέτρησης των αποτελεσμάτων μας που δεν θα είχαμε καταφέρει διαφορετικά. Ε, για παράδειγμα, ε, σενάρια, εναλλακτικά σενάρια, ε, την ανάστηληση κόστους φέλους και άλλες τέτοιες μεθοδολογίες πολύ χρήσιμες. Συλλέξαμε όλες τις πληροφορίες και τα διδάγματα και θα τις αξιοποιήσουμε στον, κατά τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης μας. υπήρξαν επίσης και ε, αποτελέσματα που θα, έχουν, θα παραμείνουν στο μακρό μέλλον χάρη στο Σίβητας. Μέσω του Σίβητας μπορέσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαμε διαφορετικά, πολύ γρηγορότερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο παρελθόν. Είχαμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε τρία νέα άτομα και αρκετό ε, ε, μη μόνιμο προσωπικό, αλλά ορισμένοι από αυτούς θα συνεχίσουν να εργάζονται ε, για μας και έτσι θα κρατήσουμε τις ε, εμπειρίες τους, δημιουργήθηκε ένα νέο, μια, ένα νέο τμήμα ε, έρευνας και ανάπτυξης που θα εστιάσει στην καινοτομία και γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο Σίβητας δημιούργησε μια θετική δυναμική στην πόλη μας. Ήταν σημαντική ευκαιρία για εμάς για να μάθουμε, για να εξελιχθούμε και για πολλούς ανθρώπους ε, αυτού μου συμπεριλαμβανομένου ήταν μια εμπειρία ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ και θα, με χαρά θα απαντήσω στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τον αντιδήμαρχο της πόλης ε, του Βίλνιους. Τα ε, ονόματα όλο και δυσκολεύουν. Είναι ο κύριος Ρώμας Αντομαβίσιους, αν το είπα καλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα σύντομα να σας σκιαγραφίσω την κατάσταση των ε, αστικών συγκοινωνιών στην πόλη μου, το Βίλνιους, και να πω εξ αρχής ότι και εμείς είχαμε θετική εμπειρία από ανταλλαγές με ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκές ε, διασκέψεις. Αλλά ε, δεν είναι ακόμα ικανοποιητική η κατάσταση. Ε, το Βίλνιους έχει 550.000 κατοίκους, η ευρύτερη περιφέρεια 700.000, μετακινούνται κάθε μέρα. Είναι μια πόλη μεσαίου μεγέθους θα έλεγα. Οι περισσότεροι μένουν μακριά από τον τόπο εργασίας τους και ε, διανύουν μεγάλες αποστάσεις και χρησιμοποιούν την τοπική συγκοινωνία, την αστική συγκοινωνία. Είδατε την πρώτη διαφάνεια, έρχομαι στη δεύτερη. Βλέπετε εδώ που βρίσκεται γεωγραφικά το Βίλνιους και εντός του κύκλου του κόκκινου ε, ζουν 15 εκατομμύρια ακάτοικοι. Και έχουμε και πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο από τη Λιθουανία και από άλλες χώρες, τουρίστες. Τώρα σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ε, πώς συνδέεται το Κάουνας με τη Βίλνιους Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κοινά προγράμματα. Ξέρετε ότι το Βίλνιους είναι και ένα σταυροδρόμι σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και πολλών άλλων διαδρόμων ευρωπαϊκών. Είναι κόμβος λοιπόν. Μεταξύ Κάουνας και Βίλνιους μετακινούνται καθημερινά πάρα πολλοί πολίτες 25.000 με 30.000 και πάνω από 100.000 αυτοκίνητα πολλές φορές. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι και οι μελέτες δημογραφικές ότι είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση των συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα και προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Αναθέσαμε μια μελέτη που χρειάστηκε μια διετία για να ολοκληρωθεί, εν μέρη με κοινοτική χρηματοδότηση. Και εδώ βλέπετε ε, πώς έχει η κατάσταση των συγκοινωνιών, ποια είναι τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, ε, κάποια ταξί ε, που είναι συλλογικά, ιδιωτικά λεωφορεία επίσης και τρία δρομολόγια τρένων που ανήκουν στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών. Αυτό είναι ο χάρτης που δεν τον βλέπετε πολύ καλά όμω, αλλά δείχνει το σύστημα ότι χωλαίνει και θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα, σε αυτή τη διαφάνεια διαπιστώνετε τις αλλαγές που έχουν γίνει στις ροές ε, της κυκλοφορίας στο Βίλνιους. 22% αλλαγή ε, σε σχέση με τις συνήθειες ε, κατά 1000% έχει αυξηθεί ε, ο αριθμός των αυτοκινήτων και 50% αριθμός των πολιτών που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση και η συμφόρηση και τα μποτιλιαρίσματα. 600 ε, αυτοκίνητα ανά χίλιους κατοίκους έχουμε και ε, δύο φορές ε, αυξήθηκε από τη δεκαετία του, μάλλον διπλασιάστηκε από τη δεκαετία του 80. Τι μας λέγουν λοιπόν οι κάτοικοι του Βίλνιους, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αποστάσεις ανάμεσα σε κάθε στάση λεωφορείου και είναι πολύ χαμηλή συχνότητα ε, των μέσων ε, ε, μαζικής μεταφοράς και είναι και σε πολύ κακή κατάσταση τα ίδια τα μέσα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε πώς έχει αλλάξει η κατάσταση και ποια μέσα χρησιμοποιούν οι επιβάτες και ποιες αλλαγές έχουν γίνει τελευταία. Δεν θα ε, μπω σε λεπτομέρειες ε, ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Βλέπετε ποια είναι τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Έχουμε ε, λεωφορεία και τρόλεϊ ηλικίας μέχρι και 30 ετών. Εκεί είναι προφανές ότι η κατάσταση στον τομέα των δημοσίων ε, μεταφόρων ε, επιδεινώνεται, διότι η χρηματοδότηση ε, δεν είναι αηφόρος και μόνιμη. Βασικός πόρος των συγκοινωνιών, 45% είναι πωλήσει συζητηρίων. Και το υπόλοιπο καλύπτεται από το Δήμο. Υπάρχουν όμως και ευνοϊκές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα μειωμένα εισιτήρια για πολύ κόσμο. Σε τι συμπεράσματα λοιπόν καταλήγει η μελέτη. Για να αλλάξει η κατάσταση και να αντιστραφεί αυτή η τάση που παρατηρείται, χρειάζονται ουσιαστικές και διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, χρειάζεται να βρούμε ένα νέο τρόπο ε, να μεταφέρουμε μεγάλο αριθμό επιβατών στους βασικούς ε, αστικούς άξονες. Στη συνέχεια θα σας αναφέρω τις λύσεις που προτείνονται. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ε, χαράξουμε ξανά ε, τις μεταφορές στο κέντρο της πόλης, νέους χώρους στάθμευσης να δημιουργήσουμε για να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το δίκτυο. Βασίζουμε τη δράση μας στις συστάσεις ε, της ε, Λευκής Βίβλου για να μειωθεί ε, η ρήπανση και να βελτιωθεί το περιβάλλον. Η μελέτη αυτή έγινε από επιστήμονες Λιθουανούς και Βρετανούς το 2010. Διοργανώσαμε μια μεγάλη διάσκεψη με εργαστήρια που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και την παρουσία εμπειρογνωμόνων από πολλές πόλεις. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τώρα ε, τα διάφορα μέσα μεταφοράς που προσφέρονται καλύτερα για την πόλη του Βίλνιους, δεδομένης ε, της ιστορίας και των υποδομών του. Σκεφτόμαστε ε, μοντέρνο σύγχρονο τραμ σιδηρόδρομο ηλεκτρικό και άλλους ε, τρόπους και άλλα μέσα μεταφόρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε ε, σε τρία είδη τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και ε, σπαστά λεωφορεία. Και καταλήξαμε στην εταιρεία Φιλέας από την Ολλανδία. Τα γνωρίζετε αυτά. Είναι προφανές ότι στο Βίλνιους χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη του κέντρου Εκεί είναι πιο μεγάλη η κυκλοφορία και η συμφόρηση και η πυκνότητα και ε, γύρω από το κέντρο όλοι οι υπόλοιποι άξονες είναι συμπληρωματικοί για να ε, υπάρχει η τοπική κυκλοφορία. Βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, στη φωτογραφία καλύτερα, πώς θα πρέπει να έχει το σύστημα αστικών συγκοινωνιών. Αυτές είναι οι συστάσεις που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, πρόκειται και για ένα νέο μέσο μεταφοράς που πρέπει να δημιουργηθεί και συστήματα με στάθμευση ε, για μετεπιβίβαση σε λεωφορείο, ε, ποδήλατα και άλλους τρόπους αηφόρας κινητικότητας. Ε, εδώ είναι η νέα χάραξη λοιπόν για την πρώτη φάση του νέου προγράμματος. Στη δεξιά διαφάνεια βλέπετε την ανάλυση της κυκλοφορίας επιβατών και οι δύο νέες χαράξεις ε, δρόμων θα μπορούσαν να καλύπτουν τη μισή κυκλοφορία. Βεβαίως, δεν μπορούμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα ολόκληρο και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πρώτα βήματα συνδυάζουμε, συνδέουμε με έξι νέα δρομολόγια το λεωφορείο με το τρόλεϊ. Με ηλεκτρονικό εισιτήριο στις 15 Αυγούστου άρχισε να ισχύει αυτό το σύστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο, το ενιαίο εισιτήριο σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Και αυτό ε, σίγουρα θα βελτιώσει την κινητικότητα των επιβατών ε, στο Βίλνους. Επίσης, Έχουμε εφαρμόσει και ένα σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιβατών. Ανισχούμε πάρα πολύ για την κατάσταση στην παλιά πόλη και στο ιστορικό κέντρο ε, του Βίλνιους. 60.000 αυτοκίνητα ε, μπαίνουν στην παλιά πόλη κάθε μέρα και είναι ε, προστατευόμενοι από την UNESCO παγκόσμια κληρονομιά η περιοχή αυτή του ιστορικού κέντρου και η παλιά πόλη. Επίσης, βελτιώνουμε τις υποδομές των μεταφορών μας. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τα νέα έργα που έχουν γίνει, ολοκληρωθεί που είναι υποκατασκευή και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τώρα ε, το δυτικό περιφερειακό δρόμο για να μειωθεί η συμφόρηση στο κέντρο και επίσης έχουμε και ένα σύστημα σύγχρονων ε, φωτεινών σηματοδοτών για να ε, περνάνε πιο γρήγορα από το κέντρο τα αυτοκίνητα και να μειώνεται έτσι η ε, ρήπαση, να μην καθυστερούν στα φανάρια. Συμπέρασμα. Το Βίλνιους ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χρειάζεται σύγχρονο σύστημα αστικών συγκοινωνιών, καθαρό που να ε, απαντά στις προσδοκίες και στις ελπίδες των πολιτών μας, των συμπολιτών μας και είναι και προτεραιότητα ε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλουμε να μειώσουμε αυτή την αύξηση των γιοταχή, ε, να δημιουργήσουμε ποδηλατόδρομους και να έχουμε και ένα σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί την ερχόμενη άνοιξη. Επίσης θα έχουμε και ένα σύστημα νοικίασης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και αντίστοιχα θα προσαρμόσουμε και τις υποδομές μας. Ωστόσο, λόγω και των οικονομικών δυσχεριών, δεν μπορεί η πόλη του Βίλνιους να επομιστεί όλο το οικονομικό κόστος 100% από ιδίους πόρους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προτεραιότητα της δημόσιας συγκοινωνίες από το 2014 και μετά. Και θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε συστήματα στάθμευσης και μετεπιβίβασης σε λεωφορείο ή σε δημόσια συγκοινωνία περίπου 30 εκατομμύρια θα χρειαστεί η πόλη του Βίλνιους για να εφαρμόσει όλα τα έργα ε, τα οποία έχουν ε, δρομολογηθεί. Ε, είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να ακούσουμε και την εμπειρία άλλων πόλεων. Δεν θα αρχίσουμε από μηδενική βάση και θα βασιστούμε στην εμπειρία που έχουν αποκομίσει άλλες πόλεις. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you, gentlemen, for your... Ευχαριστώ κύριοι για τις παρουσιάσεις σας. Και τώρα έχω τον κύριο Ελκαντράουι, ψήρα των Ευρωβουλευτών δηλαδή. Ας ξεκινήσουμε αυτό, θα δούμε μετά πιο άλλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές μας για την παρουσία τους και την παρουσίασή τους ε, για την πολιτική κινητικότητα στις ε, πόλεις τους αντιστοίχως ε, δείχνει πραγματικά ε, με ποιο τρόπο οι πόλεις βρίσκονται σε μια δυναμική τροχιά ε, κινητικότητας με πάρα πολύ μεγάλο εξυγχρονισμό και αυτό επίσης κατά την άποψή μου δείχνει ότι δεν είναι πανάκια φυσικά, δεν υπάρχει μια μαγική λύση, χρειάζεται ένα μείγμα μέτρων διότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο κάθε φορά. και δεν υπάρχει μια απλή λύση, ε, απλώς προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πράγματα καλύτερα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για σας. Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και καιρό. Έχουμε κάνει και εκθέσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου θα κάνει πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Μία από τις ιδέες που ακούγονται είναι να δοθεί η ευρωπαϊκή ενίσχυση σε συνάρτηση με την υποβολή σχεδίου αϊφόρου κινητικότητας και βιώσιμης. Η ευρωπαϊκή υποστήριξη μπορεί ε, να λάβει πολλές μορφές. Υπάρχει οικονομική υποστήριξη με το πρόγραμμα ΣΥΒΙΤΑΣ... αλλά υπάρχει και ανταλλαγή καλών πρακτικών και καλών ιδεών. Ακόμα δεν είναι αυτό το σύστημα πάρα πολύ ολοκληρωμένο, χρειάζεται να βελτιωθεί. Και θέλω να ρωτήσω και τους τρεις σας. Τι περιμένετε εσείς από εμά και από την Ευρώπη. Και έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις ακόμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυξάνονται οι ανάγκες κινητικότητας όσο αυξάνει ο πληθυσμός και μετακινείται περισσότερο. Και πολύ συχνά ακούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο ε, να δώσουμε και κίνητρα ε, τιμολογιακά. Δηλαδή, να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των πολιτών ε, και μέσω των τιμών. Συμφωνείτε εσείς αυτό και πώς μπορεί αυτό να μεταφραστεί στην πόλη σας. Τι εννοώ, ε, μπορεί να υπάρχει φόρος, ένα τέλος συμφόρησης ας πούμε ε, είναι πιο φτηνά κάποια άλλα ε, μέσα μεταφοράς, αηφόρα σε σχέση με άλλα που ρηπαίνουν περισσότερο. Το έχετε σκεφτεί αυτό στις πόλεις σας. Και μια τελευταία ερώτηση για την επιμελητία και την εφοδιαστική. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ, γιατί στην πόλη κάπως πρέπει να φτάνουν και τα εμπορεύματα. Και αυτά πρέπει να γίνονται με βιώσιμο τρόπο. Και όλο και περισσότερα υπάρχουν ε, περιοχές της πόλης που απαγορεύεται, η κυκλοφορία κάθε οχήματος. Είναι πεζόδρομοι. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε για τη τροφοδοσία, πούμε, των καταστημάτων. Ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές για την ενημέρωση και τα παραδείγματα. Δεν κατάλαβα όμως πάρα πολύ καλά. Ε, τι θέλετε από εμά, έχετε επιθυμίες, προτάσεις για μας τους πολιτικούς ή μπορείτε να λύσετε μόνοι σας τα προβλήματα αν είχατε λεφτά. Γιατί τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ ότι εκεί χωλέν. Ε, ε, καλωσορίζω και χαιρετίζω και την Ευρωπαϊκή Ευρωμάδα Κινητικότητας και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχει να κάνει μόνο με ποδήλατα ή με ε, ε, θέματα το πεζών. Η κινητικότητα είναι δικαίωμα για όλους και ιδιαίτερα για ανθρώπους με αναπηρίες και για πιο ηλικιωμένους. Θα με ενδιέφερε να μάθω αν κάνετε ιδιαίτερε προσπάθειες ε, για να μπορούν να μετακινούνται και οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με αναπηρίες. Βεβαίω, συμφωνούμε ότι οι συγκοινωνίε θα πρέπει να είναι πιο αηφόρε, να λυπαίνουν λιγότερο, να κάνουν λιγότερο θόρυβο και ένα σωρό. Και υπάρχει και μια έκκληση για μια ηλεκτρονική ή e-mobility. Ο καθένα να γνωρίζει τα δικαιώματά του, δεν λέω, αλλά και τα καθήκοντά του. Δηλαδή και οι ποδηλάτε και οι πεζοί έχουν δικαιώματα, αλλά έχουν και υποχρεώσει που θα πρέπει να γνωρίζουν. Εμείς από πλευράς ε, των νομοθετών κάνουμε πολλά για να ε, μειωθεί η κίνηση στο εσωτερικό, στα ιστορικά κέντρα των πόλεων, να υπάρχει καλύτερη υποδομή και να βελτιωθεί και η συμπεριφορά των οδηγών. Γιατί όταν συζητούμε για το κλίμα στις πόλεις δεν εννοούμε μόνο τα αιωρούμενα σωματίδια ή το θόρυβο, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ε, οι οδηγοί των φορτηγών, πώς συμπεριφέρονται στους πεζούς ή οι ε, οδηγοί αυτοκινήτων, στους ποδηλάτες. Στη δική μου πόλη ε, θέλουν να απαγορεύσουν ε, την είσοδο στην πόλη σε κάποια οχήματα συγκεκριμένα για να περιορίσουν τη σκόνη και τα ερώμενα σωματίδια. Ελπίζω να μην ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, το θεωρώ εσφαλμένο. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση ακόμα. Ο κύριος Καρλίνη είπε ότι έχετε προγράμματα που ενισχύεται ε, την ανανέωση, λέτε, του στόλου. Και τα άλλα αυτοκίνητα τι γίνεται που αποσύρονται, τα οχήματα δηλαδή, ε, τα λεωφορεία τα δίνετε στη διπλανή πόλη για να ρηπαίνετε εκείνη περισσότερο. Και το Park and Ride, ε, αυτό πώς το ενισχύεται. Γιατί τα προγράμματα ενίσχυσης δεν είναι αιώνια, είναι περασμένα χρονικά. Μετά τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάβησα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις ε, ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Πριν κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις, να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου πόλη. 400.000 είναι οι κάτοικοι της πόλης μου. Και τις ώρες εχμής έχουμε φοβερή κυκλοφοριακή συμφόρηση και το Δημοτικό Συμβούλιο του Τάλιν προσπάθησε να εισαγάγει καινούργια μέτρα. Πριν από λίγα χρόνια αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα Park and Ride, που σημαίνει ότι στους κύριους άξονες υπήρχαν χώροι στάθμευσης ε, δωρεάν Τώρα πέρασαν τρία χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε, αλλά τελικά αυτό το σύστημα δεν δούλεψε. Γιατί όσοι δουλεύουν στις γειτονικέ εταιρείε χρησιμοποιούν ε, τους χώρους στάθμευσης για να παρκάρουν δωρεάν και οι υπόλοιποι ξεκολουθούν να παίρνουν το αυτοκίνητο για να πάνε στην πόλη. Θα ήθελα να δώσω συμβουλή στους ανθρώπους ε, εδώ του Τάλιν, του Βίλνιου, συγγνώμη, να δουν τι κάνουμε εμείς και να μην κάνουν τα ίδια πράγματα. Επίσης ε, βάλαμε λεωφορείο διάδρομους, αλλά τους χρησιμοποιούν ταξιτζίδες και, τσακώ, και τσαντίζονται οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Ε, του χρόνου θα έχουμε δωρεάν συγκοινωνίες αλλά φανταστείτε, σκεφτόμαστε μάλλον για δωρεάν συγκοινωνία, αλλά φανταστείτε αυτό να εφαρμοστεί για 400.000 κατοίκου. Τι αποτέλεσμα θα δώσει. Τώρα, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να σα βοηθήσουμε. Όλα αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια και οι δράσει είναι για μια φορά. Είναι ενδιαφέρουσε ιδέε. Αναλύσατε όμω τα κάνετε μετά από αυτά, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές, τι μπορούν να κάνουν οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά συμβούλια. Έχετε νέα προγράμματα. Πώς ε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εμπειρίες σας με πιο μόνιμο τρόπο, ας πούμε. Πώς μπορούμε και εμείς να βελτιώσουμε την νομοθεσία για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Κυρία Λίχτεμπέργκερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ε, για τις λεπτομερείς σας παρουσιάσεις. Έχουν μείνει για μένα όμως κάποια ανοιχτά ερωτήματα για την Πολόνια. Μιλήσατε για όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα. Ε, τι ποσοστό του αστικού ιστού καλύπτεται. Γιατί στη Βόρεια Ιταλία ο μέσος όρος ε, ταχύτητας είναι κάτω των 30 χιλιόμετρων γιατί συχνά μποτιλιάρισμα στην πόλη. Ε, και για την Πολόνια θα με ενδιέφερε να μάθω τι γίνεται γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία με την ατμοσφαιρική ρήπανση όπως σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Διαφαίνεται εκεί καμιά βελτίωση με μια φιλόδοξη πολιτική ε, συγκοινωνιών γιατί έχει μεγάλη σημασία. Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που οι πόλεις θα πρέπει να λάβουν ριζικά μέτρα. Ας πούμε, απαγορεύεται την Κυριακή τελείωση η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Για το Βίλνιος. Αναφερθήκατε πολύ ακροθυγός στα ποδήλατα. Ξέρω ότι κάνει κρύο στο Βίλνιος, αλλά και στο Μάλμε κάνει κρύο. Εκεί να δείτε ποδήλατα που κυκλοφορούν. Και είναι και επίπεδη η πόλη σας. Ιδεώδης λοιπόν για ποδηλασία. Γιατί όταν πήγα στο Βέλνιος είδα πάρα πολύ λίγους ποδηλάτες. Ακόμα λιγότερους από τα βουνά του Τυρόλου. Γιατί δεν το αξιοποιείτε καλύτερα. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο από τη κάτι. Υποδειγματική η στάση σας και γνωρίζω ότι όλες αυτές οι πόλεις που έχουν διανύσει αυτό το δρόμο ε, για το περιβάλλον και για τη μείωση της κυκλοφορίας, σε όλες αυτές τις πόλεις υπήρξαν τεράστιες αντιστάσεις από τον κόσμο. Εσείς πώς καταφέρατε να ξεπεράσετε πρώτον αυτές τις αντιστάσεις και δεύτερον ποιες παραμένουν και σε ποιους τομείς. Και προς τους τρεις έχω μια ερώτηση. Κάτι που δεν άκουσα ακριβώς ε, από τα όσα είπατε. Τι γίνεται με την πολεοδομία παίζουν μεγάλο ρόλο και θα πρέπει να παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά τα στοιχεία και ε, στις συγκοινωνίες γιατί ε, στη περιφέρεια των πόλεων δημιουργούνται τεράστιες πόλεις ε, που είναι μόνο κοιτώνες ας πούμε ή που έχουν μεγάλα εμπορικά κέντρα και δημιουργείται τεράστια συμφόρηση και ο κύριος Ζήλε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους για τις πόλεις τους. Ο κύριος Σαββάσας ε, μίλησε για το Τάλιν και το ίδιο ισχύει και για τη Ρήγα, την πόλη μου. Και εμείς σκεφτόμαστε την ιδέα των ε, δωρεάν δημοσίων συγκοινωνιών. Κύριε από το Βίλνιους, τι γίνεται με την ποιότητα των συγκοινωνιών, αν πραγματικά τις προσφέραμε δωρεάν. Πώς θα επηρεαζόταν η ποιότητά τους. Μια άλλη ερώτηση. Ξέρουμε ότι πολλές μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη προσπάθησαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Λονδίνου και της Στοκχόλμης. Ε, βάζοντας αυτό το τέλος συμφόρηση στο κέντρο των πόλεων. Τι σκέφτεστε για αυτή τη λύση. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν εφαρμοστέο και στο Βίλνιους. Η... Πάντως στη Ρίγα και στο Τάν δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Ο κ. Ρικέ, ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές. Είμαι δήμαρχος μιας πόλης όπου υπάρχουν ίδιες συνθήκες με αυτές που ακούσαμε. Άκουσα λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Θα προσπαθήσω να είμαι απλός και να κάνω μια ερώτηση και προς τους τρεις σας. Το πρόβλημα είναι πώς θα αποφύγουμε το γεωταχή της πόλης για τη συμφόρηση, για τη ρήπανση, για την ασφάλεια κτλ. Μήπως το πραγματικό ερώτημα είναι ότι ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε τα γεωταχή είναι να δημιουργήσουμε μέτρα τα οποία είναι αποτρεπτικά. Εν παρανθέσει, άκουσα να γίνεται λόγος πολλές φορές και θα και το ερώτημα του των χώρων στάθμευσης. Αλλά όσο περισσότερα πάρκινγκ δημιουργούμε, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα θα έχουμε, ε, θα τα ελκύουμε δηλαδή και θα έχουμε περισσότερα αγιοταχή. Το να δώσουμε εναλλακτικά μέτρα στο αυτοκίνητο είναι καλό, αλλά δεν αρκεί. Είναι ικανή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη. Γιατί ε, ο κόσμος συνεχίζει να προτιμάει το αυτοκίνητο για διάφορους λόγους, αλλά και πολιτιστικούς. Το δεύτερο είναι τα αντικίνητρα που θα δώσουμε. Το ερώτημα είναι, τι αντικίνητρα δίνουμε, τι αντικίνητρα δώσατε εσείς για τη χρήση, στη χρήση των γεωταχή σε κάθε μία από τις τρεις σας πόλεις. Επίσης, υπάρχουν πολιοδομικά μέτρα για το, τους χώρους πάρκιν ε, στις ε, πολυκατοικίες. Όταν δηλαδή φτιάχνετε ε, ένα σπίτι, ας πούμε, ή όταν χτίζετε μία πολυκατοικία, είσαστε υποχρεωμένοι να έχετε και πάρκινγκ ή το εμποδίζετε αυτό. Εμποδίζετε το, την ταυτόχρονη δημιουργία και ενός πάρκινγκ. Κύριος Ντεμπάκια, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για την ε, παρουσίασή τους και τις προτάσεις των πόλεων. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σε πολλές πόλεις γίνεται λόγος για ένα ρυθμιστικό σχέδιο, master plan ε, και ε, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντα υπόψη ε, ο τρόπος λειτουργίας της πόλης, πολεοδομία, ε, κυκλοφορία. Στις μεγάλες πόλεις είναι δύσκολο. Εγώ μένω τώρα στην Αμβέρσα, αλλά έχω σπουδάσει στη Γάνδη και είναι δύο πολύ ωραία παραδείγματα για το πώς ε, ποιο είναι το παράδειγμα προς και ποιο προς αποφυγή. Η Γάνδη τα πάει καλά, η Αμβέρσα έχει ακόμα τεράστια προβλήματα. Ακούμε πολλές φορές μεγάλα λόγια και μεγαλώστομες δηλώσει, και τα λοιπά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα για συνδυασμό των διαφόρων μέσων μεταφοράς και πώς ε, ε, μπορεί να λειτουργήσει καλά αυτό. Μια δεύτερη ερώτηση μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά έχει τη σημασία του. Σύντομα, ε, πρόσφατα συζητήσαμε τις δημόσιες συμβάσεις. Διαφέρουν ακόμα πάρα πολύ οι κανόνες από χώρα σε χώρα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής. υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και δυσκολίες. Γνωρίζω την κατάσταση στο Βέλιο σχετικά καλά και ξέρουμε και τα προβλήματα, αλλά τους άλλους δύο μιλητές θέλω να ρωτήσω ε, πώς ε, γίνεται αυτό στη χώρα τους. Ε, τι γίνεται με την προετοιμασία, με τις διαδικασίες επιλογής των διαγωνισμών και την εκτελεστική φάση των διαφόρων έργων. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα των δημοσίων συμβάσεων για να δούμε γιατί έχει έρθει η ώρα να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις από την δική μου την πλευρά. Τι είδους συνεργασία υπάρχει στο εσωτερικό μεταξύ των διαφορετικών τμήματων στα δημαρχία, στην διοίκηση των πόλεων σας δηλαδή. Ας, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ε, ένα τμήμα το οποίο ασχολείται με την εκπαίδευση και αποφασίζει να δημιουργήσει ένα νέο σχολείο. Θα συντονιστεί με το αντίστοιχο τμήμα που ασχολείται με τις μεταφορές, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί χάος όταν ανοίξει το σχολείο. Ε, τα σχολεία, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν συχνά προβλήματα στην κυκλοφορία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ως παράδειγμα το φέρνω, ως ε, μια αφορμή για να συζητήσουμε κατά πόσον υπάρχει συντονισμός στις πόλεις σας. Δεύτερον, είναι κατά πόσον υπάρχει συνεργασία με την αστυνομία, με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Θα σας δώσω ένα ε, παράδειγμα. κοινά για παράδειγμα, στο το από το οποίο κατάγομαι, να δημιουργηθούν νέε ε, κατοικίες. Και θα δημιουργηθούν επίσης και θέσει στάθμευσης. Ε, δημιούργησαν λοιπόν έναν ποδηλατόδρομο και τώρα αυτό που έχει και μία λεωφορείο λωρίδα Τώρα, και ο ποδηλατόδρομος και η λορίδα χρησιμοποιείται για παρκάρισμα. Και η... τι κάνει η αστυνομία για, την... Ε, για να προστατεύσει τελικά αυτές τις υποδομές, να προστατεύσει την... Ε, τον ποδηλατόδρομο ή τη λωρίδα την ειδική για τα λεωφορεία. Γιατί όπως ξέρουμε ο αυτοκινητιστής είναι ένα περίεργο είναι άνθρωπος πριν μπει στο αυτοκίνητό του, έτσι καλός άνθρωπος, κοινωνικός, δείχνει την κατανόηση, αλλά κάτι συμβαίνει με το που μπαίνει κανείς μέσα στο αυτοκίνητο και κάθεται πίσω από το τιμόνι, δεν ξέρω τι είναι, τι, τι μεταφυσικό πράγμα συμβαίνει, αλλά αλλάζει τελείω η συμπεριφορά του. Γίνεται ένα άλλο άνθρωπο. Και η τρίτη μου ερώτηση. Στις πόλεις τις δικές σας παραπονούνται οι αυτοκινητιστές για όποιο μέτρο και αν λάβετε. Ε, αυτό συμβαίνει και εσά ή είναι κάτι, μια ιδιαιτερότητα βρετανική. Γιατί κάθε φορά που προσπαθούμε κάτι, υπάρχουν διάφοροι αυτοκινητιστές οι οποίοι, αρχίζουν να, αρχίζουν να γκρινιάζουν και να παραπονιούνται και να διαμαρτύρονται για την καταστροφή. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καλίνη τις απαντήσεις του και μετά ο κύριος Βανσεβάνεντ και στο τέλος ο πρόσωπος του Βίλνιους. Ε, κύριε Σκαλίνη που μπορώ να προφέρω καλά το όνομά σας τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις συνολικά είναι περίπλοκες θα έλεγα και πραγματικά αγγίζουν το πρόβλημα στην ουσία του. Ένα θέμα που, που επανήλθε στις παρεμβάσεις σας ήταν το πώς διαχειριζόμαστε την πόλη. Όχι μόνο το πώς θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή την κινητικότητα και την και την κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά γενικότερα πώς διαχειριζόμαστε την πόλη μας. Επίσης, μην ξεχνάτε ποιες είναι οι τάσεις. Έτσι. Από τη μία έχουμε την οικονομική κρίση, έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμπίεση της χρήσης των οχημάτων, συμπίεση και του αριθμού των οχημάτων και από την άλλη ο κόσμος επανέρχεται στα κέντρα των πόλεων, τουλάχιστον στις δικές μας πόλεις αυτό συμβαίνει. Επομένως αυξάνεται και η κυκλοφορία των γιοταχείων στους δρόμους. Μία καλή δράση υπέρ της κινητικότητας είναι να δράσουμε σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς, να σχεδιάσουμε χωροταξικά και πολυδεμικά τις πόλεις μας σωστά. Να ξέρουμε να δράσουμε με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να βάζουμε τις κατοικίες και τα σχολεία, τα γραφεία, αυτά που, ό,τι προσφέρει ας πούμε υπηρεσίες, τα εμπορικά κέντρα, αλλού ούτω ώστε να μειωθεί η κυκλοφορία. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται πάντα, μάλλον σπάνια γίνεται στην Ιταλία και επομένως στην, στην Ιταλία συμβαίνουν, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα που σας αναφέραμε. Επίσης, για να χρησιμοποιούμε πολλαπλούς τρόπους μεταφορών, θα πρέπει να έχουμε δράσεις πολλαπλές και να έχουμε και χρήση των, του μετρό και χρήση των σιδεοδρόμων και χρήση μέσων που έχουν ε, χαμηλή επίπτωση ας πούμε, στην κυκλοφορική συμφόρηση όπως ποδηλάτα και τέτοια ή ε, το να πηγαίνουμε πεζί. Επίσης, άλλος τρόπος είναι να μειώσουμε την επίπτωση στο περιβάλλον των οχημάτων που παρόλα αυτά κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Επομένως, να βελτιώσουμε ε, το στόλο των οχημάτων. Αλλά όμω αν τα κάνουμε αυτά με αυτή την προτεραιότητα, με αυτή τη σειρά που σα ανέφερα. Επομένως, καταρχάς, η δράση α, υπέρ τη βελτίωσης των αυτοκινήτων δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχουν και τα άλλα δύο, τα προηγούμενα. Καλύτερα φυσικά να, να κυκλοφορούν οχήματα μικρότερης επίπτωση στο περιβάλλον πούμε, και στην ε, συμφόρηση παρά αυτά που επηρεάζουν περισσότερο. Ε, αφού τα κάναμε όλα τα προηγούμενα, ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε και λίγα τέτοια αυτοκίνητα και να είναι όσο τον καλύτερα. Έπειτα, τι δόσεις θα έχουμε ε, δράσεων υπέρ της μείωσης της χρήσης των γιοταχή και πρόθεσης άλλων μέσων. Ξέρετε πολύ καλά το μπαστούνι και το καρότο στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε αυτή την, αυτό το κίνητρο πούμε, και αντικίνητρο. Θα πρέπει να έχουμε ένα μείγμα δράσεων, ούτω ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δράσεις της μείωσης ε, της χρήσης των γεωταχή μέσω της πληρωμής των χωροστάθμευσης ε, και από την άλλη να έχουμε συστήματα car sharing, ε, συστήματα υπέρ της χρήσης των ε, συγκοινωνιών. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σχέση αυτών των δύο. Δηλαδή, να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και τους πόρους τους οποίους ε, δρέπουμε από τα μέτρα που χαρακτηρίζονται από τον μπαστούνι, ας πούμε, να τα χρησιμοποιήσουμε, τους πόρους αυτούς, τους χρησιμοποιήσουμε, ούτως ώστε να προωθήσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Θα πρέπει αυτό να είναι σαφές και για τον πολίτη. Ότι έχουμε και αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή και αυτές τις δύο συνιστώσεις. Επίσης, είναι σημαντική η επιμελητία, η δράση μας στην επιμελητία. Υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο εδώ. Τι γίνεται με τον επιχειρηματία που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες μεταφοράς τι γίνεται με τα κέρδη του από αυτήν την επιχειρηματική του δράση. Θα πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα την επιμελητία. Δυστυχώ πολλέ από τις ε, πειραματικές ε, δράσεις μας, πειραματικές ενέργειες, δεν δώσανε θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά το όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα και που χρησιμοποιείται στην πόλη της Μπολόνιας, στο κέντρο της Μπολόνιας, που είναι τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όλοι κυκλοφορούν με 30 χιλιόμετρα ως μέγιστο όριο. Όμως και στις, στους χώρους, στις συνοικίες που είναι κυρίως, που δεν υπάρχουν γραφεία, που είναι συνοικίες, απλώς και εκεί θα πρέπει να υπάρχει όριο ταχύτητας χαμηλό, ούτως ώστε να βελτιώνει τη ζωή στη συνοικία να μην μπορούμε να ξεπεράσουμε τα 30 χιλιόμετρα. Να βάλουμε και διαφορετικά μέτρα ε, που δεν θα μας επιτρέπουν να περάσουμε 30 χιλιόμετρα, όχι μόνο να ελέγχουμε το όριο ταχύτητας. Τώρα για τις αστικές συγκοινωνίες, ε, ενδιαφέρον αυτό. Ε, πρέπει να συνδυάσουμε μέτρα που θα προσφέρουν μπαστούνι και θα πέφτει ε, που θα προσφέρουν μάλλον το καρότο και θα πέφτει και το μπαστούνι. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το σύστημα των μεταφορών, θα πρέπει να έχει μια διάσταση επιχειρηματικότητας. Καταλήγοντας, τελευταία παρέμβαση μιλούσε για τη δυσκολία να συνδυάσουμε και τον πολεμοτομικό σχεδιασμό και μέτρα παρέμβασης στον δρόμο. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τη δική μας πόλη, την Πολόνια, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει και ένας περιφερειακός νόμος που υποχρεώνει τους Δήμους και κοινότητα να έχουν μέτρα ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης, διαχείριση, ώστε να μην έχουμε μια απλή φυγή προ τα εμπρός ούτω ώστε δηλαδή να γίνεται σχεδιασμό, αλλά σχεδιασμό με συντονισμό, όχι σχεδιασμό άνευ, συντονισμού διαφόρων δραστηριοτήτων. Φυσικά αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα, γιατί δυστυχώ ο δρόμο είναι ένα πάντα. Και όταν έχει τι σωστέ διαστάσει, όλα πάνε καλά. Αλλά μία πόλη όπω όπως η Μπολόνια είναι δύσκολο να έχουμε στον ίδιο δρόμο και χώρους στάθμευσης και το ωραίο πεζοδρόμιο και ωραίο ποδηλατόδρομο και θαυμάσια λεωφο, ε, λεωφορείο λωρίδα και να κυκλοφορούν και τα οχήματα. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιε είναι προτεραιότητες. Να δούμε σε κάθε χώρο, σε κάθε περιοχή, ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς. Θα πρέπει να κάνουμε και να προωθούμε προγράμματα υπέρ αυτή τη μεταφορά και να θυσιάζουμε τι υπόλοιπε μεταφορέ, του υπόλοιπου τρόπου μεταφορά. Δυστυχώ. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε όλους τους τρόπους μεταφορών ταυτόχρονα. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ο κύριος Βανσέβενα, πολλές ερωτήσεις θα απαντήσω στα δικά μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ε, πρώτη ερώτηση. Τι περιμένουμε από την Ευρώπη. Δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Η ανταλλαγή εμπειριών το ένα και εδώ το ΣΥΒΙΤΑΣ είναι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα γιατί πέρα από την ίδια σου τη χώρα και τη βοήθεια υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια και μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες. Είναι πολύ καλά οργανωμένο και θα πρέπει να συνεχιστεί. Και το δεύτερο, ας είμαστε ειλικρινεί, βεβαίω, επιδοτήσει υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν τι πόλει για να κάνουν περισσότερα πράγματα χωρί το ΣΥΒΙΤΑΣ και χωρίς αυτά τα προγράμματα και τα μέσα, εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε στην Γάνδη αυτά που κάναμε. Βοηθάει πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, κοιτάξτε, ε, μπορείτε να μας χρηματοδοτήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάνει τα διαφορά καθημερινά. Ε, για αντικίνητρα ε, τιμών. Εμείς έχουμε 250.000 κατοίκους. Το μεγαλύτερο αντικίνητρο είναι η τιμή ε, της ε, στάθμευσης. Ένα σύστημα σαν το Λονδίνο και τη Στοκχόλμη, νομίζω η πόλη μας είναι πολύ μικρή τουλάχιστον σήμερα για ένα τέλος συμφόρησης. Για την επιμελητία και τη τροφοδοσία, το Σίβητας, ακριβώς οργανώσαμε μια πλατφόρμα συζήτησης με όλους τους ενεχομένους φορείς και ε, δίνουμε συνέχεια τώρα σε αυτή την πλατφόρμα και προβληματιζόμαστε να δούμε πώς μπορεί να γίνει ε, ας πούμε τροφοδοσία των καταστημάτων από το ποτάμι. Ε, το έχουμε δει και από άλλες πόλεις, από την Ουτρέχτη ας πούμε, και να υπάρχουν μικρά κέντρα διανομής στην περιφέρεια της πόλης και να πηγαίνουν με ηλεκτρικό όχημα στο κέντρο στα μαγαζιά. το θέμα να έχουμε ένα ειδικό σύστημα για ε, να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν προβλήματα κινητικότητας, ε, Έχουμε τέτοια προγράμματα με ειδικά ταξί. Και έχετε δίκιο και οι πεζοί και οι ποδηλάτες έχουν και δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τη συμπεριφορά ορισμένων ποδηλατών. Ρωτήσατε για τις αντιστάσεις, αν υπήρξαν και ποιες. Πριν από 15 χρόνια στη χώρα μας, ε, πεζοδρομήσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή ε, και ενημερώσαμε τους πάντες. Ε, είπαμε ποια θα είναι τα πλέον ε, το κοινό πληροφορήθηκε, αντίδρασαν κυρίως οι έμποροι που δεν πίστευαν ότι θα λειτουργήσει αυτό. Ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσεις τις αντιστάσεις είναι να υλοποιήσεις το έργο και μετά να δείξεις τα πλεονεκτήματα για να πιστούν και οι υπόλοιποι. Εγκρίνιαξαν λίγο τώρα πριν από 15 χρόνια έγινε αυτό και τα τελευταία δέκα χρόνια δεν αμφισβητεί κανείς ε, τους πεζοδρόμους. Είναι φανταστική η κατάσταση και ο τουρισμός πάει πολύ καλά και το εμπόριο θαυμάσια. Κανείς δεν θυμάται πώς ήταν πριν ούτε ζητάει να γίνει. Βεβαίως η χωροταξία και η πολεοδομία είναι σημαντική και τι κάνουμε. Ε, όταν κάνουμε το σχέδιο κινητικότητα συνεργαζόμαστε και με του πολεοδόμου, αυτού που φτιάχνουν το ρυθμιστικό σχέδιο ε, και κάνουμε αυτή τη συνεργασία και ανταλλαγή είναι απαραίτητο, αλλιώς δεν λειτουργεί η κατάσταση. Κάτι άλλο που με ρωτήσατε για τις δωρεάν συγκοινωνίες στην πόλη μας έχουμε, αλλά για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Ε, τα παιδιά 6 με 14 ετών για να μάθουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ε, ως συγκοινωνιολόγος το ξέρω αυτό ότι πρέπει ε, όμως να ε, υπάρχει και ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι στην πόλη Χάσελτ ήταν τελείως ε, δωρεάν οι συγκοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα τριπλασίασαν όμως και τη δυνατότητα μεταφοράς. Ε, ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε για αποθάρρυνση. Σας είπα, το σημαντικότερο είναι η στάθμευση. Τα τελευταία 15 χρόνια στο εσωτερικό της πόλης, στο ιστορικό κέντρο, δεν ε, ε, φτιάχτηκε κανένα πάρκινγκ. Έχουμε υπόγεια γκαράζ 600 ε, ας πούμε 600 θέσεις όταν χτίζεται ένα υπόγειο γαράζ όμως 600 θέσεων καταργείται ένα επίγειο 600 θέσεων δεν δημιουργούνται νέες θέσεις παρκαρίσματος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αντικίνητρο και σε συνδυασμό με τη σωστή τιμολόγηση με βάση την αγορά. Δηλαδή να μην είναι ε, κάτι που συμφέρει να κατεβαίνει ε, ο άλλος με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης και να δουλεύει όλη μέρα και να πληρώνει το, το πάρκινγκ. Και επίσης οι κατοικίες... Ε, ε, όταν χτίζονται κατοικίε, βεβαίω προβλέπεται στάθμευση, γιατί πού θα το βάλει το αυτοκίνητο άλλο στο δρόμο. Με τα γραφεία είναι άλλη η κατάσταση και ο σχεδιασμό. Μπορούμε να εγκρίνουμε στο κέντρο ορισμένες, όμως πολύ περιορισμένες σε αριθμό θέσεις στάθμευσης για τα γραφή. Ε, τι γίνεται με τις συνδυασμένες μεταφορές. Ε, κλασικό παράδειγμα είναι το Park and Ride για μετεπιβίβαση. Ε, και με το Civitas όμως έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια Park and Bike. Δηλαδή αφήνεις το αυτοκίνητο σου και παίρνεις ποδήλατο. Φτάνει στην άκρη της πόλης, ας πούμε, και μετά παίρνεις ένα μικρό ποδήλατο και κυκλοφορείς στην πόλη. Προσπαθούμε να το προωθήσουμε αυτό Ε, και στο Park Ride δίπλα να υπάρχουν χώροι που να νοικιάζουν ποδήλατα. Υπάρχουν δυνατότητες και μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες, όχι μόνο αυτές. Άλλο, αυτό που ρώτησε ο Πρόεδρος, συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών. Βεβαίως συνεργάζονται οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και η επιθεώρηση για τα σχολεία, η... όταν χτίζεται ένα σχολείο ή όταν χτίζεται ένα εκθεσιακό κέντρο. Βεβαίως συζητούμε και με τους πολεοδόμους γιατί μας αφορά αυτό. Εκ των προτέρων, αν μπορούμε να εκτιμήσουμε αν είναι καλή τοποθεσία ή όχι. Αλλιώς εξεπερνούν οι εξελίξεις, τρέχεις να τις προλάβεις και η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Βεβαίως, εκ των προτέρων συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Ωραίο αυτό που ρωτήσατε ε, για τις ε, υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Έτσι, αστυνομία το λέμε αυτό εμείς απλά. Ε, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε με την αστυνομία. Εντάξει, είναι και η τροχέα. Δεν... Εντάξει, εμείς μια αστυνομία, έχουμε αστυνομία τη λέμε. Εντάξει, η αστυνομία ε, έχει συμφωνίες ε, συνάψει μαζί μας, ακριβώς για συγκεκριμένα θέματα να κάνουμε και εκστρατείες ενημέρωσης, αλλά προσπαθούμε πάλι σε συνεννόηση με την αστυνομία, όταν υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος που είναι πάντα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προσπαθούμε ε, να βάλουμε εμπόδια, κάποια κολονάκια ή ας πούμε και, και ε, τυχεία ε, για να μην μπορούν να παρκάρουν. Και βοηθάει η αστυνομία σε αυτό. Και τελευταίο, αν διαμαρτύρονται οι οδηγοί, βεβαίω και διαμαρτύρονται οι οδηγοί, παντού το ΙΟΤΑΧΗ, αλλά και οι οδηγοί έχουν και παιδιά και εγγόνια και οικογένειες και Μπορεί ε, όταν παίρνει ένα μέτρο να μην είναι 100% υπέρ του οδηγού, αλλά μπορεί να του πει είναι υπέρ των παιδιών σου και των εγγονιών σου και τότε θα το καταλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντομαβίσιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα στη, με τη σειρά με την οποία τέθηκαν. Κύριε Σκόκ, ρώτησε εάν θα ήμασταν σε θέση να λύσουμε μόνοι μας τα, ε, τα προβλήματά μας χωρίς εξωτερική βοήθεια χρηματική. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα ήμασταν σε θέση να το κάνουμε και ήθιστε τη χρηματοδότηση να συνδέεται με ορισμένα κριτήρια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Κοινοβούλιο ε, διαφέρουν από την πραγματικότητα και θα ήταν καλύτερα να έχουμε περισσότερα ε, ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά τα παλαιά τεχνολογίας ε, οχήματα. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται γιατί κανείς δεν θέλει να τα αγοράσει. Προσπαθούμε, δεν προσπαθούμε μάλλον προσπαθήσαμε να πουλήσουμε παλιά λεωφορεία μας, παλιά τεχνολογίας σε άλλες χώρες όπως το Καζακστάν και κανείς δεν ήθελε να τα αγοράσει. Μου αρέσει η ιδέα που παρουσιάσατε και συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την υλοποίηση ενός συστήματος Park and Ride. Ε, θα επισκεφτώ το Τάλιν τον Οκτώβριο ε, επισκέφτηκα και πριν 6 μήνες την ε, πόλη σας και συζητήσαμε την ε, πιθανότητα, τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα δωρεάν δίκτυο δημόσιων μεταφορών. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει μάλλον να αλλάξουμε την ορολογία και να χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις, να λέμε για παράδειγμα ότι το δωρεάν δημόσιο σύστημα συγκοινωνιών θα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν θα χρηματοδοτείται από τα εισιτήρια. Μου κίνησε το ενδιαφέρον το σύστημα αυτό που χρησιμοποιείται στο Τάλιν και άλλαξα γνώμη όταν άκουσα τα επιχείρηματά σας. Πιθανώς ένα τέτοιο σύστημα να ε, λειτουργούσε και στη δική μου πόλη και να αντιμετώπιζε προβλήματα όπως η ρήπανση και η συμφόρηση κάνοντας πιο ελκυστικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Τώρα, απευθύνομαι στο, στην εκπρόσωπο από την Λεκτονία. Εάν ε, εισαγάγουμε ένα δωρεάν σύστημα δημόσιων συγκοινωνίων δεν θα αλλάξει τίποτα και αυτό που θα χρειαστεί τελικά είναι να αλλάζουμε πιο συχνά το στόλο των οχημάτων και πού θα βρεθούν οι πηγές χρηματοδότησης ενός τέτοιου συστήματος είναι προφανές ότι τα οχήματα που κυκλοφορούν στο Βίλνιους είναι 10 και 20 ετών. Το κόστος χρήσης τους έχει αυξηθεί κατά 2,5 ε, φορές. Άρα ίσως θα έπρεπε να εισάγουμε ε, περιβαλλοντικούς φόρους ή κάτι αντίστοιχο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα έτσι ώστε να εισπράττουμε φόρους ε, από τις επιχειρήσεις στη βάση της, των μεταφορο, της μεταφοράς των εργαζομένων τους. Επομένω θα περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του συστήματος που θα κάνει το Τάλιν. Σχεδιάζουμε ε, να διεξάγουμε μια δημοσκόπηση μεταξύ των πολιτών του Βιλνίους, να τους ρωτήσουμε κατά πόσο τους ενδιαφέρει ε, κατά πόσο θα ήθελαν να έχουν ένα τέτοιο σύστημα δωρεάν μεταφορών, συγκοινωνιών. Επίσης μπορώ να πω ότι έχουμε και εμείς προβλήματα συμφόρησης και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο ε, δημιουργήσαμε τις έξι γρήγορες λεωφοριολορίδες. Υπολογίσαμε την μέση ταχύτητα και η μελέτη μας μας έδειξε ότι θα καταφέρναμε να έχουμε 25 ε, με 30 χιλιόμετρα την ώρα ε, και αυτό θα ήταν η ταχύτητα της γρήγορης λεωφοριολορίδας ε, και κάτι που θα καθιστούσε τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο ελκυστικές. Στον αφορά τα ποδήλατα, έχουμε 100 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, ενώ το συνολικό μήκος των οδών ε, είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Άρα μπορούμε να κάνουμε πολλά εδώ. Έχουμε, σχεδιά, έχουμε δημιουργήσει ένα σχέδιο για τη δημιουργία δρόμων. Πάντα φυσικά το θέμα είναι χρηματοδότηση. Τώρα στο θέμα της πολιοδομίας και της χρήσης γης. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Στο κέντρο του Βίλνιους παραμένουν ορισμένες βιομηχανικές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στην παλιά πόλη που είναι προστατευόμενη κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Επομένως πρέπει να αλλάξει η χρήση αυτών των περιοχών, να δημιουργηθούν σε αυτές τις περιοχές, να, να μετατραπούν μάλλον σε περιοχές πεζοδρομημένες. Ένα ακόμα πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει. Προσπαθούμε να ε, οι ορισμένες εταιρείες να μετα, μετεγκατασταθούν σε κατοικημένες περιοχές, κάτι που θα μας επιτρέψει να, μειώσουμε την κίνηση και τη συμφόρηση στο κέντρο της πόλης. Επίσης υπήρξε μια ερώτηση σε σχέση με τον τρόπο μείωσης του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων. Αυτό συνδέεται και με οικονομικά στοιχεία. Όταν υπολογίζουμε ότι ένα ταξίδι με το ΙΟΤΑΧΗ κοστίζει 6 φορές περισσότερο από το να χρησιμοποιηθούν τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, μεταφοράς, αυξήσαμε το κόστος στάθμευσης στο κέντρο του Βιλνίους μέχρι και τρεις φορές και όταν δημιουργούνται νέα, ε, όταν χτίζονται νέα κτίρια είναι ε, απέτηση, είναι υποχρεωτικό κάθε ε, διαμέρισμα να έχει και χώρο στάθμευσης που αντιστοιχεί σε αυτό. Στο Βίλνιους διαθέτουμε 10, 10 υπαίθριους χώρους στάθμευσης που ε, στους οποίους μπορούν οι κάτοικοι να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να ε, περπατήσουν στο κέντρο. Όσον αφορά το γενικό ρυθμιστικό σχέδιο, ναι, έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο στη διευθυνσή μα και οι δημόσιες οι αποτελούν σημαντικό στοιχείο αυτού του σχεδίου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα επιτρέπαμε να κτιστεί ένα νέο σχολείο χωρίς να σχεδιαστεί πρώτα η εξυπηρέτησή του από το Δημόσιο συστημαστικών Συγκοινωνιών ως αντιδήμαρχος του Βίλνιους τα τελευταία τρία χρόνια. Γνωρίζω ότι όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ε, εάν το έργο είναι σαφές και απλό, ε, καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό μέσα σε ένα χρόνο, ενώ διαφορετικά αν είναι πιο περίπλοκο χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός με πολλά συναρμόδια υπουργεία, πρέπει να διεξάγουμε μελέτες ε, επιπτώσεων και όλες αυτές οι μελέτες, όλη αυτή η φάση διαρκεί περίπου δύο χρόνια, ενώ η φάση της υλοποίησης μπορεί να διαρκεί μόνο έξι με 8 μήνες. Και τώρα όσον αφορά τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται, οι κάτοικοι, οι περίοικοι του ε, κέντρου ε, διαμαρτύρονται για εκείνους που έρχονται από, ε, εκτός του κέντρου, από τις, τα προάστια και έρχονται να εργαστούν στο κέντρο. Αλλά προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις μετακινήσεις των πολιτών μελετήσαμε την πιθανότητα να ε, δημιουργηθούν νέα δρομολόγια. Και η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν υπέρ της επέκτασης του δικτύου των δημοσίων συγκοινωνιών. Ε, Αλλά η πλειονότητα των πολιτών στο Βιλνίους χρησιμοποιεί το γιοταχή τους. Εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία λοιπόν. Πάντα λέμε στους πολίτες μας ότι από τη στιγμή που κάποιο ζει σε μία πόλη, ε, συστηματικά και συνέχεια κάνει συμβιβασμού σε όλα τα επίπεδα. Ε, στην τομέα της δημόσια υγεία, στην τομέα της ρήπανση, στην τομέα του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, ομιλητές μας και τον κύριο Καλίνη και τον κύριο Βανσέβεναντ και τον κύριο Δωμαβίσιους για τη σημερινή σας έλευση και συνεισφορά και τις απαντήσεις. Ε, ευχαριστώ και την Αντιπρόεδρο Τυρό για την εισαγωγή της. Είναι επίκαιρη, όπως είπαμε, μια ακρόαση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κινητικότητας και ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακούσαμε τις εμπειρίες των τριών πόλεων σας ε, που είναι τελείως διαφορετικές και από διαφορετικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε και για τους βουλευτές πρέπει να πω ότι έχουμε ένα τέταρτο διάλειμμα και μετά κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ.